Okay, it seems that we can start now. Good afternoon. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Καλωσορίζουμε τα, τους νεοεκλογέντες. Ε, συγχαρητήρια και στους προηγούμενους συναδέλφους, τους οποίους αναγνωρίζω εδώ, τους παλαιότερους συναδέλφους. Μου ζητήθηκε να προεδρεύσω στην αρχή της συνεδρίασης σήμερα, διότι είμαι από ό,τι φαίνεται δυστυχώς η πιο παλαιά ε, το πιο παλαιό μέλος, εκεί, εδώ. Οπότε προεδρεύω. Ε, θυμίζω λίγο τους κανόνες ε, στους συναδέλφους. Θέλουμε σήμερα να ε, ορίσουμε το Προεδρείο, να εκλέξουμε το Προεδρείο της Επιτροπής και τους Αντιπροέδρους με βάση το άθρα 2 και 3 τον, του εθνικού κανονισμού. Η σύνθεση του Προεδρείου λοιπόν θα πρέπει να αποτυπώνει την ποικιλομορφία ε, του Κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά ε, άντρες ή γυναίκες και δεν μπορεί να προέρχονται από τα ίδια κράτη-μέλη. Ερχόμαστε τώρα στις εκλογές. Όπως είπα, πρώτα εκλέγουμε τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπροέδρους. Θα ήθελα για άλλη μια φορά, με βάση τους κανόνες, ε, να ανακοινώσω τα ονόματα των αναπληρωματικών μελών που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, διότι δεν υπάρχει ε, απαρτία. Ο κ. Άντζελ Τζαμπάσκι, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κυριάκο Βελόπουλο, η κυρία Μαραβιτσότο θα αντικαταστήσει την κυρία Τζάντσα, ο Άνταμ Κόζα την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για το ΕΛΚ, ο Σβέν Σούλ θα αντικαταστήσει τον Λορόν Τζόρτζι Βίντσε της ΕΛΚ, από το ΕΛΚ για άλλη μια φορά, και ο Δημήτρης Παπαδάκης αντικαθιστά τον Άλφρετ Σαντ της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Υπάρχει κάποιος άλλος που αντικαθιστά κάποιο μόνιμο μέλος, κάποιο τακτικό μέλος, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ο ομιλητής. εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια και δεν μπορούμε να μεταφράσουμε. Μάλιστα, σημειώθηκε λέει η πρόεδρος, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημειώθηκε. Ναι, θα προσπαθήσω να αντικαταστήσω τον κύριο Μπερέγκλιο. Δεν είμαι βέβαιος ότι καταφέρω. Could you say again the name of the, of the member that you are replacing, please? Ποιον αντικαθιστάτε, είπατε. Μπορείτε να μας ξαναπείτε. Δεν άκουσα το όνομα. Ποιον αντικαθιστάτε. Είμαι ο Ρίτσαρ Κόρμπετ και με ποιον Σμερίλιο. Σμερίλιο είναι το όνομα του βουλευτή που αντικαθιστώ. Ναι, Κρίστιαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την κυρία Ευρέν από το ΕΛΚ. Okay, nobody else it seems. Yes, you may be needing your card. Ναι, ενδεχομένως να χρειαστείτε την κάρτα σας. Ωραία. Θα περάσουμε τώρα στην εκλογή του Προέδρου. Θα πρέπει πρώτα να δούμε αν υπάρχει απαρτία. Νομίζω ότι υπάρχει. Χρειαζόμαστε νέα μέλη. Δεν χρειάζεται νομίζω να μετρήσουμε. Νέα μέλη υπάρχουν σίγουρα. Και τώρα οι υποψήφοι στην Προεδρία ε, θα πάρουν το λόγο. Yes, you have the floor. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι. Okay. Frau Vorsitzende, wir schlagen für den... Κυρία Πρόεδρε, προτείνουμε την κυρία Μονσεράτ για Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. Thank you. Do we have any... Ευχαριστώ. Άλλοι υποψήφοι υπάρχουν. We don't. We then have only... Μάλλον δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Ένας υποψήφιος για την θέση του Προέδρου, λοιπόν, η κυρία Μονσεράτητα, είστε εδώ. Ε, συμφωνείτε να λάβετε την Προεδρία. Ωραία, ευχαριστώ. Ε, τώρα πρέπει βεβαίως να επιβεβαιώσω ότι είστε τακτικό μέλλον. Είστε, μέλος, είστε τακτικό μέλος. Έχετε συμπληρώσει τη δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα. Το ίδιο ισχύει και τη δήλωση για τον κώδικα συμπεριφοράς. Ναι, μπορούμε λοιπόν να σας εκλέξουμε διαβοής για χειροκροτήματος. Toutes mes félicitations et je vous propose d'échanger nos places. Συγχαρητήρια, μπορείτε να πάρετε θέση. Τη θέση μου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να προέδρω αυτή τη σημαντική επιτροπή. Αυτή η επιτροπή είναι η πόρτα εισόδου για του Ευρωπαίου πολίτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία στην επόμενη θητεία να ακούσουμε, να φουγκραστούμε τα προβλήματα των συμπολιτών μα να τους βοηθήσουμε να τα επιλύσουν. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να φέρουμε το Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Εγώ θα είμαι δίκαιη, θα σεβαστώ το κράτος δικαίου. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με όλες τις πολιτικές ομάδες, επικοδομητικά και υπεύθυνα για να υπερασπιστούμε το συμφέρον των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Και τώρα, αν μου το επιτρέπετε, θα μιλήσω αυτή την υπέροχη γλώσσα, τα ισπανικά. Πρώτα απ' όλα, ε, έχουν προβλεφθεί, ανέφερε η Πρόεδρος προηγουμένως, ε, τα αναπληρωματικά μέλη οπότε μπορούμε να περάσουμε τώρα στην εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι υποψήφοι για αυτή τη θέση. Θα ήθελα ε, στο όνομα των Πρασίνων να προτείνω την Τατιάνα Ζδανόκα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλος? Εάν συμφωνείτε λοιπόν, μια και υπάρχει μονάχα... συγγνώμη, συγγνώμη, λησμόνησα. Η κυρία Τατιάνα Ζδανόκα. Δέχεστε να είστε αντιπρόεδρος. Oh, thank you. Ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, βεβαίω, συμφωνώ. Και έχετε ε, υπογράψει και όλες τις απαραίτητες δηλώσεις. Άψογα και τέλεια. Άρα έχουν καλυφθεί οι προϋποθέσεις και μια και έχουμε μονάχα μία υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία, την πρώτη αντιπροεδρία της Επιτροπής αυτής, εάν συμφωνείτε, ε, διαβοής ε, να εκλέξουμε και την ε, συνάδελφο και παρακαλώ ελάτε εδώ στο Προεδρείο δίπλα μου να καθίσετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα. Μάλλον όχι. Το ΕΛΚ ζητά το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ δύο λεπτά διάλειμμα λόγω της ε, αλλαγής της ε, σειράς στα ονόματα. Θέλω να διαβουλευτώ με την πολιτική μου ομάδα σχετικά με τους υποψήφιους για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Δύο λεπτά διάλειμμα ζητώ. Δύο λεπτά μόνο. Πρόεδρος, εάν συμφωνείτε ε, οι υπόλοιπες ομάδες, μια και μία ομάδα ζητά ε, ε, παύση δύο λεπτών. Παρακαλώ να γίνει δεκτό το αίτημά του. Σταματούμε λοιπόν για δύο λεπτά. Sí, apreciados miembros. Αγαπητοί συνάδελφοι, παραπάνω από δύο λεπτά έπερασαν. Επομένως, να ξαναρχίσουμε. Θέλει να πάρει το λόγο κάποιος εκπρόσωπος πολιτικής ομάδας. Ελκα. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι παρούσα σήμερα η πολιτική μου ομάδα για να ψηφίσουμε πρόεδρο και αντιπρόεδρους και ε, είχαμε μία συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων αλλά βλέπουμε τώρα ότι δεν τηρείται αυστηρά η συμφωνία αυτή και γι' αυτό πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη διαβούλευσης ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και γι' αυτό ζητάμε αναβολή της ψηφοφορίας. Los no. Perfecto. Sí, Ο κύριος Παπαδάκη. Εμείς ε, εισηγούμαστε να συνεχίσει κανονικά η, η διαδικασία και να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία για κάθε θέση ξεχωριστά. Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, το ΕΛΚ λοιπόν έχει ζητήσει, έχει έχει ε, πάνω από 7 ε, βουλευτές ε, έτσι ώστε που συμφωνούν ας πούμε με την αναβολή της ψηφοφορίας. Η σοσιαλιστική ομάδα αντιτίθεται, επομένως πρέπει να ψηφίσουμε για το κατά πόσον θα αναβληθεί η συνεδρίαση. Επομένως, με το πράσινο κουμπί Λοιπόν, πράσινο σημαίνει ότι είμαστε, είναι κάποιος υπέρ της αναβολής, ενώ με το κόκκινο θα ψηφίσει αυτός που θέλει να συνεχιστεί η ψηφοφορία. Πριν όμως θα δώσω το λόγο στον κύριο Γάνιας. Θέλω να αναγγείλω, κυρία ε, Πρόεδρε, ότι η κυρία Βομβίσε δεν είναι εδώ και την αντικαθιστώ εγώ. Ε, empezaríamos um, la votación y la vamos Ωραία, πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν. Perfecto. Nadie me ha pedido, <laughs> si no secreto no, Επομένως, ε, νομίζω δεν υπάρχει λόγος ε, να ψηφίσουμε μυστικά, να ψηφίσουμε διανατάσεως της χειρός. Υπέρ της αναβολής της συνεδρίας της Επιτροπής. Υπέρ της αναβολής. si les parece, como desde también los servicios técnicos ah, Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι επειδή έχει πρόβλημα και η τεχνική υπηρεσία εδώ να καταγράψει τους, ε, τις ψήφους, ε, να ξεκινήσουμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω ότι όσοι ψηφίσουν με το πράσινο κουμπί θέλουν την αναβολή, όσοι ψηφίσουν με το κόκκινο θέλουν να, διακοπ... θέλουν να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. De 30, de 30 votaciones. Ψηφίσαντες 30, 18 κατά τις αναβολές και 12 υπέρ. Άρα συνεχίζουμε την ψηφοφορία περνάμε στην ψηφοφορία, του, στην εκλογή μάλλον του δεύτερου ε, αντιπροέδρου του Προεδρείου. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, παρουσιάσω την υποβάλω την κυρία Λιάννα Τόμ ε, από την ομάδα Renew Europe. Κάποια άλλη υποψηφιότητα. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Α, ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Μιούλερ θέλει να πάρει το λόγο. Okay. Um, acepta Δέχεστε να είστε δεύτερη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών. Yes, thank you. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ και να σας πω ότι έχω ήδη υπογράψει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχει άλλη ε, υποψηφιότητα, διαβοής. Και σας παρακαλώ και εσάς να έρθετε εδώ. Continuamos. Ωραία, τώρα είμαστε στον τρίτο αντιπρόεδρο. Έχει κάποια ομάδα να προτείνει υποψηφιότητα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ECR θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Ρίτσαρτ σαρνέσκι ως τρίτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Ήδη έχει υπηρετήσει στην Επιτροπή αυτή σε μια από τις προηγούμενες θητείες. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Δεύτερη αντιπρόεδρος θέλει το λόγο. Λάθος κουμπί πατάω μάλλον. Ε, δεν έχω να προτείνω αλλά εκ μέρους ε, της ομάδας Renew Europe ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να, να ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία. Αυτή είναι η πρόταση της Renew Europe. Ε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, χρειάζομαστε υποστήριξη αυτής της πρότασής σας από 7 μέλη Πόσα μέλη λοιπόν υποστηρίζουν αυτήν την πρόταση, έτσι ώστε ενδεχομένως να γίνει αποδεκτή. Sí, sí, levante la mano quien apoye hacer la votación en secreto. Ok. Sí, ok. Como se cumplimenta el requisito. Ωραία. Καλύφθηκε αυτή η προϋπόθεση των 7 συμφωνούντων άρα να ψηφίσουμε με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πριν από αυτό όμως, για την θέση της τρίτης αντιπροεδρίας υπάρχει άλλος υποψήφιος όχι. Επαναλαμβάνω ότι με το πράσινο ψηφίζουμε υπέρ του υποψηφίου, με κόκκινο ε, κατά ε, του υποψηφίου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν άρχεται. όμως. Λοιπόν, 31 ψηφίσαντες, 18 υπέρ του κυρίου Τσερνέσκη, 10 κατά και 3 αποχέ. Και επομένως εξελέγει ο τρίτος αντιπρόεδρος κ. Στερνέτσκι ε, και παρακαλώ ελάτε εδώ να καταλάβετε την θέση που σας αρμόζει και σας αντιστοιχεί. Si, si les parece, Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην τελευταία τέταρτη αντιπροεδρία, τέταρτος αντιπρόεδρος. Έχετε προτάσεις? Παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών προτείνουμε την Κριστίνα Μαέστρε, Κριστίν Μάκρο, την κυρία που κάθεται δίπλα μου. Άλλες υποψηφιότητες. Όχι, επομένως διαβοής νομίζω ότι μπορούμε να την εκλέξουμε. Συγχαρητήρια. Φαντάζομαι ότι ήδη έχετε υπογράψει τα, τις απαραίτητες δηλώσεις και φαντάζομαι επίσης ότι δέχεστε αυτήν την θέση. Ωραία λοιπόν. Παρακαλώ να καθίσετε. Uh, Ενημερώνω τους συναδέλφους ότι έχετε πρόσβαση πλέον στην εφαρμογή που είναι η βάση δεδομένων όπου ε, καταγράφονται οι αναφορές και όλες οι σχετικές πληροφορίες. Εάν ένας ε, βουλευτής θέλει να έχει πρόσβαση και ο βοηθός του σε αυτή την εφαρμογή πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα. Θα λάβετε μια επιστολή άλλωστε με όλες τις λεπτομέρειες. Θα... Επίσης έχουν μοιραστεί οι θηρίδες, ε, στις θηρίδες ε, το κείμενο με τις αναφορές, ε, για την ώρα μόνο στα αγγλικά, μεταφράζεται και σε άλλες γλώσσες όμως. Και εφόσον έχουμε εκλέξει τα μέλη του Προεδρείου, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συνεδρία, θα τα ξαναπούμε 4 και 5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους και ευχαριστώ πολύ.